may ask you to take seat. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε με την ακρόασή μας. Θα ήθελα όσοι παρευρίσκεστε να, να κάθεστε στις θέσεις σας, όχι σε θέση άλλων και μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακρόαση από την αίθουσα ακρόασης και μέσω της ε, ιστοσελίδες μας και μόνο τα μέλη μπορούν να χειροκροτούν. Καλημέρα σας. Η κυρία Ολσφογκ είναι πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και ο κύριος Μπούζεκ από την Επιτροπή ε, Ενέργειας, Έρευνας και Περιβάλλοντας και εγώ από την Επιτροπή ΕΚΟΝ θα ήθελα να καλωσορίσουμε τον κύριο Κατάινεν ο οποίος ε, είναι υπεύθυνος ή θα είναι υπεύθυνος για την απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα. Εάν λοιπόν και επειδή το χαρτοφυλάκιο ε, σχετίζεται με την εργασία των ε, επιτροπών αυτών, ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη τους. Επίσης, ε, εμπλεκόμενες επιτροπές είναι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Μεταφορών. Συνεπώς, θέλουμε οι επιτροπές να κρίνουν κατά πόσο ο υποψήφιος επίτροπος μπορεί να είναι μέλος του διευθυντηρίου και να αναλάβει το εν λόγω χαρτοφυλάκιο. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι πριν από την ακρόαση ο υποψήφιος επίτροπος απάντησε γραπτό σε ένα ερωτηματολόγιο το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί σε όλες τις κοινοτικές ε, ε, γλώσσες και επίσης έχει υποβάλει και μία δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Η Επιτροπή Γιούρη δεν έχει παρατηρήσει ως προς τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων του υποψηφίου επιτρόπου. Ο υποψήφιος επίτροπος θα προβεί σε μία εισήγηση 15 λεπτών και στη συνέχεια θα, έχουμε 5, θα διαθέτει μάλλον 5 λεπτά για μία καταλεκτική δήλωση. Μετά θα υποβληθούν 45 ερωτήσεις από τους ε, Ευρωβουλευτές. Ένα λεπτό η ερώτηση και δύο λεπτά η απάντηση από τον υποψήφιο επίτροπο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ευρωβουλευτές ότι η αρχή των τριών λεπτών θα εφαρμοστεί αυστηρά. Υπάρχει διερμηνία σε 23 γλώσσες, άρα όλοι οι ομιλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μητρική τους γλώσσα. Και μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακρόαση από την ιστοσελίδα μας. Ως πρόεδρος ΣΥΚΟΝ θα ήθελα να κάνω ορισμένα εισαγωγικά σχόλια θα πρέπει η νέα Επιτροπή να φτάσει σε φιλόδοξους στόχους μέσα στα πλαίσια της ανάκαμψης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της όθησης της εργασίας στην πραγματική οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη και την κρίση που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια. Άρα το πακέτο των 300 δις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούγκερ για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις ε, σχετίζεται με το όλο θέμα και θα ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, όπως αναφέρεται στην ε, επιστολή, αφορά την, ε, τις υποδομές, έρευνα, καινοτομία και υποδομές, έτσι ώστε οι άνεργοι να επανέλθουν στην αγορά εργασίας με αξιοπρεπή εργασία. Επίσης, με την εγγύηση για τους νέους θα πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους και ε, τη χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων τους. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συντονίσουν αυτές τις δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τη, τον κοινωνικό αντίκτυπο της διαρθρωτικής ε, μεταρρύθμισης μετά την απόφαση των συντονιστών της Επιτροπής ΕΚΟΝ ε, ζήτησα περαιτέρω διασαφήσεις από τον πρόεδρο Γιούγκερ σε σχέση με τον επιμερισμό ευθυνών στον οικονομικό τομέα σε σχέση, και ιδιαίτερα σε σχέση με την εξωτερική και εσωτερική εκπροσώπηση της Επιτροπής και αναμένουμε τις απαντήσεις του ε, Προέδρου. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαρίτα Ούσεμπογκ. Ευχαριστώ, θα μιλήσω στα Σουηδικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στον οικονομικό τομέα. Έχει μεγάλη σημασία να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση για να προωθήσουμε όμως αυτές τις ε, δραστηριότητες, δεν θα πρέπει να υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός και θα πρέπει οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι να την χάνουν προστασίας. Μία πραγματική αγορά δεν θα πρέπει να ε, συρρυκνώνει την αγορά και τις συλλογικέ συμβάσεις. Δεν θα πρέπει να υπάρχει συρρύκνωση ή παλινοδία και ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών ε, μελών, διότι υπ' αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων και να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά, να λειτουργήσει σωστά η αγορά εργασίας. Επίσης, οι ιδιαίτερα χαμηλοί μισθοί δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Βλέπουμε ότι ανακύπτει εθνικισμός και λαϊκισμός, όλο ένα και περισσότερο. Γι' αυτό κύριε Κατάινεν, είναι πολύ σημαντική η θέση σας και το χαρτοφυλάκιό σας. Άρα η λέξη απασχόληση είναι πολύ σημαντική μέσα στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου σας. Ευχαριστούμε την κυρία Μαρίτα ε, Ουλσκοκ και τον κύριο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Σας ευχαριστώ που συμπροεδρεύετε σε αυτή την ακρόαση είναι η τελευταία μέρα των ακροάσεων και αυτό είναι ένα καλό νέο για τους ευρωβουλευτές. Παρευρεθήκαμε σε πολλές ακροάσεις. Έγιναν πολλές συζητήσεις για τα ευρωπαϊκά ε, θέματα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Γιούρκη Κατάινεν που ε, είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος για τη νέα Επιτροπή και να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους από την ε, ΕΚΟΝ, την Επιτροπή Απασχόλησης και ε, όλους τους εκπρόσωπους των ΜΚΟ, ΜΜΕ, ΜΜΕ βιομηχανίες και κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια δημόσια ακρόαση την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν οι πάντες. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακρόαση στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω και εγώ ορισμένα λόγια για τη δική μου επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την έρευνα, καινοτομία, ε, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ, ενέργεια, ψηφιακή οικονομία. Όλα αυτά τα, όλες αυτές οι συνιστώσεις ε, προωθούν την ανταγωνιστικότητα και εμπίπτουν στους τομείς ε, του υποψηφίου επιτρόπου, που θα πρέπει να συντονίσει και με άλλους επιτρόπους. Μέσα στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου του έχουμε πολλές προκλήσεις για την επόμενη πενταετία σε όλους αυτούς τους τομείς και οι συνάδελφοι από την Ήτρε, την οποία εκπροσωπώ, θέλουν να γνωρίσουν πόσο ο υποψήφιος επίτροπος προτίθεται να ανταποκριθεί. Δηλαδή να ανταποκριθεί στις ε, προσδοκίες των ε, πολιτών. Θα ήθελα τώρα ο κύριος Γκουαλτιέρη να αναλάβει την ακρόαση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ. Ο κύριος Κριστιανής Χάρινς έχει το λόγο. Δεν είναι σκόπιμο να ακούσουμε πρώτα τον Επίτροπο. The introductory remarks were very interesting and but very quick but... Ναι, ναι, ναι. Ας ακούσουμε και την εισήγηση. Έκανα, ε, έκανα λάθος. Ε, μετά την πέμπτη